Καλημέρα συνάδελφοι. Πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι το σύστημα παρουσίασης ηλεκτρονικών το ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίασης αποτελεσμάτων έχει βλάβει. Άρα δηλαδή, ίσως να μην βλέπουμε πάρα αυτά τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να τα διαβάζω. Ξαναξεκινάω λοιπόν, το ξαναλέω. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίαση αποτελεσμάτων μπορεί να έχει κάποια βλάβη, που σημαίνει που σημαίνει ότι ε, θα βλέπετε μόνο κάποια στοιχεία από την ψηφορία και όχι το αποτέλεσμα. Κατόπιν, όσον αφορά την προστασία των ζώων, εκεί ψηφίζουμε για την σύσταση και τη δεύτερη ανάγνωση ε, προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Συνάδελφοι, με βάση το άρθρο 165 του Κοινοβουλίου ζητώ να αναπεμφθεί το θέμα στην Επιτροπή. Για πάρα πολλά χρόνια ε, παρακολουθήσαμε αυτή την οδηγία και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία τροποποιούνται σημαντικά ε, και πρέπει να γίνει αυτό για να υπάρχει προστασία των ζώων. Η έγκριση αυτή τη ε, νομοθεσία θα επιτρέπει τα πειράματα για διδακτικού σκοπού και την χρησιμοποίηση πολλέ φορέ του ίδιου του ζώου που θα του προκαλεί πόνο. Θα πρέπει λοιπόν να στηθούν άλλε εναλλακτικέ λύσει. Το θέμα δεν είναι να καταλήξουμε σε μια ακραία θέση, αλλά να σεβαστούμε το άρθρο 13 τη Συμφωνία που αφορά στην λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα λαμβάνεται πλήρω υπόψη η ευζοία, η καλή κατάσταση των ζώων. Δεν θέλουμε να αναχαιτήσουμε την έρευνα, κάθε άλλο να την ενθαρρύνουμε. Είναι λοιπόν απαράδεκτο να λέμε ότι θα εγκρίνουμε αυτή την οδηγία για να την τροποποιήσουμε κατά επόμενα έτη. Α αναλάβουμε λοιπόν την ευθύνη που μα. Ε, αρμόζει, που μας προσήκει. Δεν είναι πολιτική ή ιδεολογική η απόφαση, είναι θέμα ε, λογικής και η λογική μπορεί να έχει και πολιτικό χρώμα. Mrs. Πρόεδρος, κύριε Αλφάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για την πρότασή σας. Έχουμε 40 συναδέλφους που θέλουν να σηκωθούν και να στηρίξουν αυτή την πρόταση. Μπορείτε να σηκωθείτε παρακαλώ. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε τους 40 ε, συναδέλφους και τώρα ε, ένας ε, υπέρ της πρότασης. Νομίζω η κυρία Evans είναι πρόθυμη να στηρίξει αυτή την πρόταση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα μας ε, στηρίζει την αναπομπή γιατί και εμείς ε, έχουμε πολλές επιφυλάξεις για το κείμενο ΣΕΧΗ. Τώρα πλέον τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας των ζώων. Αλλά αυτή η νέα νομοθεσία θα το εμποδίζει αυτό στο μέλλον. Άρα δηλαδή δεν θα υπάρξει βελτίωση και αυτό είναι κατά αυτού που συμφώνησε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Επίσης ε, πρέπει να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι οφείλουμε να αναζητούμε ένα εναλλακτικά μέτρα εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Επίση πρέπει να υπάρχει σαφέστατο ορισμό των προποθέσεων ε, για την ε, χρήση ε, μη ανθρώπινων όντων Υπάρχουν διαφορετικέ ευερμηνίε από αυτού στα κράτη-μέλη. Πρέπει να γίνει και άλλη συζήτηση για το θέμα και γι' αυτό και για άλλα θέματα για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει απόλυτη σαφήνεια και επίση και το ότι η νομοθεσία αυτή θα είναι αποτελεσματική. Ε, κατά ο κύριος Δεκάστρο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ω ε, πρόεδρο τη ε, Επιτροπή Γεωργία που είναι αρμόδια, εγώ είμαι κατά τη ε, αναπομπή στην Επιτροπή. Διότι διάρκεισε η συζήτηση 1,5 χρόνο και εκεί εκφραστήκαμε ξεκάθαρα υπέρ τη συμβαστική πρόταση που επιτεύχθηκε και δεν τοποθετήκε κανεί αρνητικά. Μόνο δύο αποχέ. Άρα δηλαδή δεν βλέπω κανένα λόγο να επανεξεταστεί το κείμενο. Υπάρχουν σήμερα όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνηγορούν μπορούν στο να ψηφίσουμε σήμερα. Η κυρία Γίγκλη, η παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ομολογώ εκπλήσωμε με την πρόταση της ε, συναδέλφου. Σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια η συνάδελφος δεν ήταν καν παρούσα όταν συζητήθηκε το θέμα. Εκπλήσωμε ε, με αυτή την πρόταση της κυρίας Ιβάνς ε, ε, της σκιώδης των Πρασίνων ήταν παρούσα σε όλες τις τριμερείς συζητήσεις και σε 7 Απριλίου όταν καταλήξαμε σε συμφωνία συμφώνησε. Οι Πράσινοι κατέθεσαν τροπολογίες στην Επιτροπή Γεωργίας που θα καταθέσουν εκ νέου σήμερα. Αυτό βέβαια είναι νόμιμο και περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε σήμερα. Ε, εσείς ε, λοιπόν ακούσατε ότι όλες αυτές οι τροπολογίες απορρίφθηκαν από τις υπόλοιπες ε, πολιτικές μας εκτός των πρασίνων. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι σας παρακαλώ θερμότατα με αυτή τη συμβαστική πρόταση που ούτε και εγώ συμφωνώ απόλυτα και νομίζω κανείς δεν υπάρχει εδώ στην που μπορεί να είναι ικανοποιημένος απόλυτα με αυτή τη συμβαστική πρόταση. Σας παρακαλώ όμως παρόλα αυτά να εγκρίνουμε αυτή τη συμβαστική πρόταση, να απορρίψουμε την προφορική πρόταση που κατέθηκε γιατί αλλιώς θα έχουμε την παλιά οδηγία του 86 και με αυτήν θα αναγκαστούμε να συνεχίσουμε να ζούμε όσον αφορά τα πειράματα στα ζώα. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε τώρα ένα βήμα προς την κατεύθυνση της καλύτερης προστασίας των ζώων. Σας ευχαριστώ. Διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να διευκνήσω λιγάκι τη θέση της πολιτικής μου ομάδας και να πω ότι μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να ε, παρακολουθεί κανείς ως πολιτική ομάδα μια τριμερή συζήτηση. Όταν διαπιστώνουμε ότι η συγγήτρια δεν θέλει να συνειδητοποιήσει ότι ο αριθμός ε, των πειραμάτων σε ζώα με βάση αυτόν τον κανονισμό θα αυξηθεί, ο αριθμός των πρωτογενών πειραμάτων και αυτός θα αυξηθεί και τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβούν σε αυστηρότερα μέτρα, ε, τότε νομίζω ότι έχει κανείς δικαίωμα να προτείνει την αναπομπή στην Επιτροπή. Και αν δεν γίνει δυνατό κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί σωστά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Well, thank, thank you for illuminating your group's... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εξηγήσατε τις δυσκολίες της πολιτικής σας ομάδας όσον αφορά το θέμα αυτό. Νομίζω ότι όμως το σώμα είναι κυρίαρχο και θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Όσοι λοιπόν είναι υπέρ της πρότασης για να πούμε στην Επιτροπή, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι. Όσοι είναι υπέρ. Κατά. Συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Ε, απορρίφθηκε η πρόταση. Το πρώτο λοιπόν θέμα είναι το πρώτο θέμα με ονομαστική ψηφορία, άρχεται η ψηφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μπορούμε να δούμε τους αριθμούς, άρα δουλεύει το σύστημα. Ε, η τροπολογία υπερθμών 2 με ονομαστική ψηφορία άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε, ψηφίσαμε. Και αυτή απορρίφθηκε. Πάμε στην τροπολογία 3, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία και αυτή απορρίφθηκε. Έτσι λοιπόν εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γίγκλε. Πάμε τώρα στην έκθεση ΕΡΙ, κατευθυντήριες γραμμές. Ο κύριος Ντάβιτ έχει το λόγο για διαδικαστικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Τι τελευταίε δύο μέρε πήραμε 400 mail για το θέμα αυτό. Θα μπορούν οι υπηρεσίε σα κάτι να κάνουν για να μην περνάμε και εμεί το χρόνο μα ε, και διαγράφοντα τα μηνύματα. Κοιτάξτε, στο Outlook, ε, στο computer σας μπορείτε να πατήσετε ένα κουμπί και να σβήσετε αυτόματα όλα τα μηνύματα, αλλά βέβαια εντάξει αυτό είναι θέμα που αφορά εσάς και τους ε, ψηφοφόρους σας. Ε, επίσης διαδικαστικό. Είναι τραγικό αυτό που είπατε. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι ψηφοφόροι σα να έρχονται σε επαφή μαζί σας. Αν εσεί δεν το θέλετε, μα ποιο τελικά είστε. Thank you for amplifying my Ευχαριστούμε πολύ που ενισχύσατε και στηρίξατε αυτό που είπα, αγαπητοί συνάδελφε. Πάμε τώρα σε 32 τροπολογίες από την Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, ψηφίζουμε ε, ενσώματη, με ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Το αποτέλεσμα το βλέπετε στην οθόνη. Πάμε τώρα σε μια σειρά τροπολογιών. Δεν με ακούτε? Ε, θα μιλάω πιο δυνατά. Τροπολογία 5. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 13. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 16. Παρακαλώ ε, σηκώστε το χέρι Είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται ε, αποχές εγκρίνεται. Η 19 ονομαστική ψηφορία, συγγνώμη, ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 28 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και αυτή εγκρίνεται. 30 με ονομαστική ψηφορία. Ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία και αυτή εγκρίθηκε. Πάμε στην 40. Υπέρ παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 55 με ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 31. Ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 η τροπολογία με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίθηκε. Η 52 υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Η 53 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Η 9 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 60 με ονομαστική ψηφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 61 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφορία παρακαλώ. Έκλεισε. Και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 54. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 62 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 63 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Επίσης εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση που τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματο ε, ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται με ευρία ψηφία. Συγχαρητήρια. Κύριε Αβελή. Επόμενο σημείο. Επτά σχέδια ψηφίσματο. Και ένα διαδικαστικό. Det gäller ändringsförslag 48 och det har insmugit sig ett fel när det gäller... Πρόεδρε, στην τοπολογία 38 υπάρχει ένα σφάλμα. Ιδίω στην σουηδική μετάφραση. Μιλάμε για ελάχιστο μισθό και ελάχιστο εισόδημα. Οι μεταφραστικέ υπηρεσίε παρακαλώ να κάνουν την ανάλογη διόρθωση. Σα ευχαριστούμε κύριε Λούινσον. Οι υπηρεσίε θα προχωρήσουν στην διόρθωση. Και άλλο διαδικαστικό. Θα ήθελα να παρακαλέσουμε το Συμβούλιο να δεχθεί ε, την ψηφοφορία, το πετρέλαιο της ψηφοφορίας και να τοποθετηθεί σήμερα, τώρα. Also ich den Rat auf, unserer Stellungnahme zu folgen. Thank you. In fact... Καλό το Συμβούλιο να δεχθεί τη θέση. Το Συμβούλιο παρέστη στην συζήτηση. Άκουσα το όσα είπαμε και προφανώ θα λάβει υπόψη σοβαρά τα όσα είπε το Κοινοβούλιο, όπω μα είπαν και χθε το βράδυ ο κ. Μπουτικόφερ. Θέλετε το λόγο. Εγώ με το μηχάνημά μου μπορώ να υπερψηφίζω και όχι να καταψηφίζω κάτι που με τρομοκρατεί. Τι είναι αυτό. <laughs> In the immortal words, we'll send a technician. Όπως λέμε και στον κόσμο των θνητών, θα σας στείλουμε ένα τεχνικό. Και τώρα, για τα ψηφίσματα. Πρώτα απ' όλα, κοινή η πρόταση ψηφίσματος. Κύριε Μάρο, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, επειδή στον κατάλογο ψηφοφοριών μου δεν βλέπω την αίτηση για ονομαστική ψηφοφορία, και επειδή είναι τόσο σημαντικό το θέμα και υπάρχει και ανάλογη συμφωνία με των ομάδων, θα έλεγα να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία την ε, τελική πρόταση ψηφίσματο. Το σημειώνω. Ο κύριο Χάουιτ. Εγώ έμαθα, πρόεδρε, ότι υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία για τι τροπολογίε και με τη δική σα διακριτική ευχαίρεια ζητώ να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση. Δεν υπάρχουν τροπολογίε. Όμω την κοινή πρόταση ψηφίσματο θα την ψηφίσουμε χωρί να έχω αντίρρηση για ονομαστική ψηφοφορία. Όμω θέλω να μάθω εάν υπάρχουν αντιρρήσει από άλλου συναδέλφου. Αν 40 έχουν αντίρρηση, δεν μπορεί να γίνει. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσει, ψηφίζουμε την πρόταση. Με συγχωρείτε. Κύριε Χάουιτ, θέλετε ξεχωριστές ψηφοφορίες για τις, για παραγραφούς, δηλαδή να ψηφίσουμε για τις καταγελαμένες ήδη ψηφοφορίες. Με νομαστική ψηφοφορία τα πάντα δηλαδή. Μάλιστα. Παράγραφος 7. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Σωστή παρατήρηση. Ο κύριος λέει ότι δεν θέλει ονομαστική ψηφοφορία για τι επιμέρου παραγράφου, αλλά μόνο για το τελικό κείμενο. Είναι λογική ε, άποψη. Τώρα ψηφίσουμε την παράγραφο 7. τα ισχυρό. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Αιτιολογική σκέψη 5. Και τώρα κοινή πρόταση ψηφίσματο. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 658 υπέρ, 1 κατά 22 εποχές. Πολύ σαφές το μήνυμα νομίζω. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Yes. Ένα διαδικαστικό της κυρίας Ντεκάιζερ. Ήθελα να ψηφίσω και το μήνυμά μου νομίζω ότι έχει καταγραφεί και να καταγραφεί και στα πρακτικά παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε. Okay. Thank you so much. Right, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει και την οικονομική παράλληλη πρόοδο. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε σκοπιμότερε